και το κοινό τόσο πολύ παρακολουθεί εδώ πέρα την συζήτησή μας. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίες συνεδρίας και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται.